Pronti, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σε όλους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε ψηφοφορίες. Οπότε λάβετε θέσεις. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, εγκρίνεται η μερίζια διάταξη. Για τεχνικούς λόγους σας ενημερώνω ότι η διερμηνία δεν μπορεί να υπάρχει σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής μας σήμερα. Οι, χώρες, οι γλώσσες που λείπουν είναι τα βουλγαρικά, τα δανικά, τα ουγγρικά, τα λιθονικά και τα σλοβενικά. Να σας πω ότι η σημερινή συνεδρίαση αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο. Και τώρα ξεκινάμε με το σημείο 3 της σημερινής διάταξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε τώρα για το δικό μου σχέδιο έκθεσης για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2003-17 του Συμβουλίου δεδομένου ότι η Κομισιόν δεν έχει ευθυγραμμίσει τις ε, παλαιές διατάξεις επιτροπολογίας στο σύστημα των ε, κατά εξουσιοδότηση πράξεων, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη. Έχω προτείνει μόνο δύο επιτροπολογίες που αφορούν την επιτροπολογία. Ωστόσο, όπως είχα ανακοινώσει στην τελευταία μας συνεδρίαση, θα ήθελα να υποβάλω και μια προφορική τροπολογία για λόγους ε, νομικής ε, νομικού τύπου. Πρόκειται για μόνο ένα εκτιμώντας, ε, το οποίο επεξηγεί τις άλλες δύο Τροπολογίες, ότι δηλαδή τα άρθρα της Παλαιάς Επιτροπολογίας θα πρέπει να διαγραφούν, διότι αυτή τη στιγμή είναι ασύμβατα με το σύστημα των κατεξουδότηση πράξεων που εισάγονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και ειδού το κείμενο, και θα σας το διαβάσω στα αγγλικά. Πρόκειται για το εκτιμώντας 4α νέο. Οι διατάξει της απόφασης 2003 κάθετος 17 κάθετος Ευρωπαϊκή Κοινότητα που παραπέμπει στην απόφαση του Συμβουλίου τη 28 Ιουνίου 1999 ε, ε, παρουσιάζουν τις διαδικασίες για την άσκηση εφαρμοστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται στην Κομισιόν θα καθυστερηθεί γιατί η εφαρμογή του στο πλαίσιο αυτή της απόφασης θα ήταν ασύμβατη με το σύστημα των κατεξοδότηση και πράξεων και εφαρμοστικών αρμοδιοτήτων που εισάγονται με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης της Λισαβόνας αντιστοίχως. Αυτή είναι η προφορική ε, τροπολογία. Αν συμφωνείτε μπορούμε τώρα να περάσουμε στη ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ, συμφωνείτε όλοι, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία διανατάσεις της χειρός. Ποιοι είναι υπέρ κατά, άποχες, ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία η προφορική που μόλις σας διάβασα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία επί του κειμένου όπως τροποποιήθηκε, ποιοι είναι υπέρ, κατά κατά αποχές κανείς ωραία σας ευχαριστώ και περνάμε στο σημείο 4 σημείο 4 όπου έχουμε κάποια προβλήματα και θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Άλπερτ Ντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο μέλλον θα κάνω μια τροπολογία, ίσως και σήμερα να την κάνω και να ζητήσω. Ε, να μην ψηφίζουμε κείμενα που παραβιάζουν το άρθρο 146 παράγραφος 1. Θα πρέπει όλα τα γραπτά κείμενα του Κοινοβουλίου να υπάρχουν στις επίσημες γλώσσες. Δεν επιτρέπεται να έχουμε τροπολογίες εδώ και μάλιστα και συμβιβαστικές μόνο στα αγγλικά παραβιάζεται εδώ ο κανονισμός του Κοινοβουλίου τα δικαιώματα των βουλευτών και δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να ψηφίζω ε, κείμενα που δεν είναι στις επίσημες γλώσσες, γι' αυτό ζητώ τώρα αναβολή της ψηφοφορίας. Ehm, Ευχαριστώ, Άλμπερτ. Έχεις απόλυτο δίκιο, Άλμπερτ Σύμφωνα με τον κανονισμό, όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες. Να, σίγουρα το λέει αυτό ο κανονισμός, δεν υπάρχει αμφιβολία όμως. Λαμβάνοντας υπόψη την ε, ε, ελαστικότητα με την οποία αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα στο παρελθόν σε πολλές ε, περιπτώσεις, θα σας πρότεινα, αλλά φυσικά θα δεχτώ τη γνώμη της πλειοψηφίας, θα πρότεινα λοιπόν για σήμερα Αν συμφωνείτε να κάνουμε όπως και κάναμε και στο παρελθόν, αλλά να πούμε στην γραμματεία ότι από σήμερα και στο εξής για σημαντικά κείμενα όπως για παράδειγμα η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, όπου προφανώς εκεί μιλάμε για νομοθετικές εκθέσεις τεράστιας σημασίας, να προχωρήσουμε με βάση τον κανονισμό, άρα να μεταφράζονται τα κείμενα σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης. Βεβαίως, αυτή η απόφαση που θα λάβουμε σήμερα, πέρα από το γεγονός του αν θα ψηφίσουμε ή όχι την έκθεση του Γουφσκι, θα αλλάξει και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες για την ψηφοφορία, για το φάκελο ε, μεταρρύθμισης τη κοινή γεωργική πολιτική μέχρι τον Νοέμβριο, όπω είχαμε σκεφτεί, εν πάση περιπτώσει για την συνεδρίασή μας του Δεκεμβρίου. Ε, θα δυσκολέψει πάρα πολύ λοιπόν αν, όπως σας προτείνω, εφαρμόσουμε αυτόν τον κανόνα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το λάβουμε υπόψη, ότι δηλαδή θα καθυστερήσουμε. Γιατί η μετάφραση των τροπολογιών σε όλες τις γλώσσες καθιστά απαραίτητη παίρνει χρόνο, τουλάχιστον δύο-τρεις εβδομάδες παραπάνω. Συμφωνείτε όλοι να ψηφίσουμε σήμερα και να ξεκινήσουμε με αυτή την πιο περιοριστική ερμηνεία από την προηγούμενη φορά ή θέλετε να αναβάλουμε την ψηφοφορία της έκθεσης Φωσιγόφσκι που... Ε, θα ψηφίσουμε λοιπόν. Ε, ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Δέσ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σωστά ε, έθεσες το ζήτημα και το ερώτημα αν συμφωνούν όλοι. Γιατί αρκεί και να διαφωνεί ε, ένας και μόνο συνάδελφος ή μία συνάδελφος δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεσμεύεται από τον κανονισμό η διαδικασία. Γι' αυτό σήμερα... Εντάξει, είμαι διατεθειμένος να το αποσύρω, αλλά στο εξή, αν δεν υπάρχουν σε όλε τι επίσημε γλώσσε τα έγγραφα, δεν πρόκειται να δεχτώ ψηφοφορία. Grazie Albert. Ha chiesto la parola Martin Ευχαριστώ, Μάρτιν Όσλινγκ, ζήτησε το λόγο. Ε, ο κύριος Χόισλινγκ, έχει ε, τυπικά απολύτω δίκιο ο Άλβερτ. Ισχύει αυτό από τον κανονισμό, αλλά τα δύο πράγματα που πρέπει σήμερα να ψηφίσουμε, οι προθεσμίε ήταν τόσο σφιχτέ και τόσο μικρέ. προσπαθήσαμε μέχρι τέλο και για την έκθεσή μου για τα αντιβιωτικά να καταλήξουμε σε συμβιβασμού. Δεν υπάρχει θέμα κακής βούλησης εδώ. Είναι χρονικό και μόνο. Ε, παράλληλα γίνονται και οι διαπραγματεύσεις ε, για την ΚΑΠ και δεν είναι απλό. Θα παρακαλούσα και θα χαιρόμουν να ψηφίσουμε σήμερα και τις δύο εκθέσεις αν γίνεται για να ε, τηρήσουμε τουλάχιστον τις προθεσμίες και την επόμενη φορά όταν θα έχουμε τέτοιο θέμα στην ημέρησια διάταξη συμφωνώ απολύτως. Αλλά τώρα πραγματικά πιεζόμαστε πάρα πολύ από το χρόνο. Bene, e ευχαριστώ τον Μάρτιν Ευχαριστώ και τον Άλμπερ Ντες. Αν συμφωνείτε λοιπόν όλοι, θα προψηφίσουμε τώρα όπως προβλεπόταν και να πούμε στη γραμματεία αυτό το θέμα, ότι δηλαδή δεν θα απομακρυνθούμε από, τις, από τους κανόνες της επόμενης ψηφορίας. Άλμπερτ και πάλι έχει το λόγο. Ναι. Το δικό μου παράπονο έχει σχέση με το εξής. Δεν μπορούμε όλα να τα περνάμε με τέτοιους ρυθμούς του σκοτωμού σε σημαντικά θέματα τέτοια που αφορούν 27 κράτη-μέλη, μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους, με την ησυχία μας να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε σωστά τα θέματα. Γιατί εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να υποστώ τις συνέπειες όταν έρθουν να μου τις καταλογίσουν τι είναι αυτά που ψηφίσατε. Γιατί στο παρελθόν επανειλημμένα το έχουμε ζήσει αυτό. Ευχαριστώ, Άλμπερτ. Ποιο ζήτησε το λόγο, ο Άγνιου. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προβάλλω ένσταση για αυτή τη διαδικασία, δηλαδή πρέπει να ακολουθούμε και εμείς τους δικούς μας κανόνες αν πρόκειται να νομοθετήσουμε και να ρυθμίσουμε πράγματα άλλων. Vabbè, siamo tutti d'accordo. Grazie anche di quest'ultimo intervento. Ripeto per chiarezza, όχι, ωραία. Ε, ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία με αυτήν την ε, ε, ελαστικότητα. Να ψηφίσουμε. Από τις επόμενες ψηφοφορίες θα σεβαστούμε τον κανονισμό. Και φυσικά θα πρέπει και να δεχτούμε τις επιπτώσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία... Για να τάσω τη θα έχουμε πολλέ ψηφοφορίε, γι' αυτό θα προσπαθήσω να προχωρήσω όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί είναι γεμάτη η μέρα μα και πρέπει να κάνουμε και συνεδρίαση των συντονιστών στο τέλο. Allora dobbiamo procedere con la voto elettronico. Avete tutti la scheda dentro? Έχετε τι κάρτε σα για να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάμε λοιπόν. Συμβιβαστική 3. Α, όχι, όχι, όχι. Άρθρο 1. 68. Ε, Ντελάνζε. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έχουμε τους, δημοκρατι... Ε, τους σοσιαλίστες, έχουμε έναν παραπανίσιο στους σοσιαλιστές, συγγνώμη. Ε, συμβιβαστική τρία. Συμβαστική τρία. ψηφίζουμε. Chiusa la votazione. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγινέται. Transport 3. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται θα έλεγα. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Συμβιβαστική 4. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. pagina successiva, emendamento 79, aperta la votazione. Τροπολογία 79. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Ψηφίζουμε όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 88 τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία NV18. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Έγκρινεται. Συμβιβαστική 6. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Η 6 λοιπόν εγκρίνεται. Περνάμε στη 235 τώρα. Εράντς Γκαρσία και άλλων. Ψηφίζουμε. Ε, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εκρίνεται και η συμβαστική 8. Στην επόμενη σελίδα περνάμε και ψηφίζουμε την τροπολογία 58. 58. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Τροπολογία 58. Έγκρινεται. Τροπολογία 65. Επόμενη. Κάντεμπαχ και άλλοι. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Τροπολογία 75, 65 απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την NV7. NV7 Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρανς 5. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Envy 27 ψηφίζουμε τώρα. Ένβη 27. Τέλος ψηφοφορία απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Πρώτο τμήμα. Προσέξτε λίγο παρακαλώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κατά τμήματα ψηφοφορία στις συμβιβαστικές. Εδώ όμως κάνουμε μια εξαίρεση και σε αυτή την περίπτωση προσοχή για τις επόμενες φορές και το λέω για τις ομάδες. Συμβιβαστική 9 πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα της συμβαστικής 9. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής έννεα. το οποίο αντιθέτως απορρίπτεται τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προχωράμε. Τροπολογία 160. 160. Όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. Όχι στην 160, πάμε στην επόμενη σελίδα που είναι η 182 Delange. Μάλιστα. Ψηφίζουμε τροπολογία 182. Chiedo un attimo al segretariato, un momento. Μισό λεπτό ρωτάω τη γραμματεία. momento, eh, perché col fatto dello split vote c'è un'interpretazione. Μισό λεπτό γιατί με τη χωριστή ψηφοφορία πρέπει να δούμε τι πρέπει ακόμα να ψηφίσουμε. Ok, allora un attimo di attenzione. Dobbiamo votare l'emendamento 162 Πατράων Εβές. Ναι, πρέπει να ψηφίσουμε την 162 Πατράων Εβές. 162. Ψηφίζουμε. Περνάμε και ψηφίσουμε για την 163. 163 είναι η επόμενη. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 165. Είναι η ίδια πλειοψηφία, προβλέπω. Απορρίπτεται όντως. 166. 166. Η ίδια πλειοψηφία. Απορρίπτεται. 164. Ψηφίζετε όλοι. Απορρίπτεται. 168 τώρα. Εγκρίνεται. Πάμε στην επόμενη σελίδα τώρα. Στην 171. Μάνερ. 171. Απορρίπτεται. 172. Ψηφίζουμε. Votazione chiusa. Εγκρίνεται. 173. Ψηφίζουμε. Votazione chiusa, direi 170. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 174. Ψηφίζουμε για την 174. Ταραμπέλα. Votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 175 άλβες. Εγκρίνεται. Με 176. Votazione aperta. Votazione chiusa. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Τρανς 5. Απορρίπτεται. Εκατόν εβδομήντα εφτά. έγκλε. Εγκρίνεται. 181 Άλβες. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 18 προς 20. 182 Ντελάνγκε. Stazione chiusa, direi in questo caso approvato. Εγκρίνεται. Και τώρα συμβιβαστική 10. Συμβιβαστική 10 ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Πάμε στην. Ε, εγκρίνεται και πάμε στην 192, Νεντελτσέβα. 192. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, απορρίπτεται. 193. Πόλσεν και άλλοι. Αν 194 τελάγγε. 194 τελάγγε. Ψηφίσατε όλοι. Έγκρινεται. 195 ψηφίζουμε. Τέλος πληροφορίες. Απορρίπτεται. Τώρα... Εκατόν ενενήντα Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Πάμε στην ε, τροπολογία της Επιτροπής Μεταφορών. Τραν 6. Εγκρίνεται και πάμε στην βεστική 11. Ο εισηγητής θέλει το λόγο. Prego. Il relatore ha chiesto la parola. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δημιουργείται πρόβλημα με την έλλειψη μετάφρασης. Ε, πίστευα ότι θα είχαμε αρκετό χρόνο, αλλά δεν είχαμε. Θα ήθελα για την τροπολογία 11 να προσθέσω, να καταθέσω μάλλον μια προφορική τροπολογία. Ε, αναφερόμαστε στη μεταφορά των ε, αλόγων και 12 ώρες είναι η ανώτατη προθεσμία για να μεταφερθούν στα σφαγεία. Μπορώ να σας το διαβάσω στα αγγλικά, αν θέλετε. Ε, παρά τις νέες επιστημονικές, ε, τα νέα επιστημονικά τεκμηρία σε σχέση με τις προθεσμίες μεταφοράς ε, των λοιπόν από τον Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων, βάσει του οποίου συστήνεται κατανότατο όριο ταξίδι 12 ώρων, δεν συμπεριλήφθησαν σχετικές συστάσεις για αλλαγές στην νομοθεσία μέσα στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει συντομότερο χρόνο μεταφοράς για όλες τις μετακινήσεις σε τα σφαγεία βάσει του κανονισμού 2009-156 βάσει των ε, επιστημονικών ε, στοιχείων της ΕΦΣΑ και βάσει και της ε, γραπτής δήλωσης του Κοινοβουλίου ε, της 25 Φεβρουαρίου 2012. Πάντως μιλάμε για τις 12 ώρες διότι αυτή είναι η σύσταση ε, της ΕΦΣΑ και μιλώ συγκεκριμένα για τα άλογα γιατί δεν ισχύουν για τα υπόλοιπα ζώα οι ίδιες ανώτατες προθεσμίες. se ci sono obiezioni o Τώρα πρέπει να ρωτήσω αν κανείς είναι αντίθετος με την πρόταση της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Ωραία λοιπόν. Ψηφίζουμε. Προχωράμε. Συμβιβαστική 11. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Συμβιβαστική 11. Προσοχή. Βλέπω πως τώρα ψηφίσατε όλοι και απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την επόμενη. 202 ψηφίζουμε. Όχι. Όχι. Συμβιβαστική και την ψηφίσαμε και απορρίφθηκε. Ε, λοιπόν, ψηφίσουμε την ε, συμβιβαστική 11 χωρίς την προφορική ε, τροπολογία. Συμβιβαστική 11, λοιπόν, γίνεται δεκτή. Η 11 λοιπόν η συμβαστική γίνεται δεκτή, αλλά η προφορική τροπολογία επ' αυτής όχι. Ωραία, πάμε στην ε, ε τροπολογία 1. Στην ενοποιημένη λοιπόν τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Συμβιβαστική 12. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάμε στην επόμενη σελίδα, στη 219. Τροπολογία 219 θα λέγω ότι απορρίπτεται. ΕΝΒΙ NV3. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται ναι, όχι. Ναι. 19-19. Ισοψηφία, αλλά απορρίπτεται. Έμβη 26. Η... αρχή Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 26. «234. Στρίφλερ υπέρ, ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία, τέλος της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 1 της Επιτροπής Μεταφορών, δεύτερο τμήμα, ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τραν 10 τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας. Θα λέγα ότι εγκρίνεται. 245 Σμιτ. Εγκρίνεται. ΕΝΒ22 τμήμα 2. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Σωστά, δίκιο είχα να απορρίπτεται. 247. Τροπολογία 247, Κάντεν και άλλοι. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Όχι, εγκρίνεται. Εγκρίνεται 247 και πάμε τώρα στη 248. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προτελευταία. NV21. Τέλος της ψηφοφορίας. Αγνιού. Μα ψηφι... με δουλεύουν ολονών τα μηχανήματα. Τι θέλετε να ξανακάνουμε την ψηφοφορία για την NV21. Ωραία. Ας ξαναψηφίσουμε. NV21. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ε, ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 τώρα. Εγκρίνεται. 232. 232 στρίφλερ. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην 261 γέγκλε. 261. Και άλλες ψηφοφορίες. Ε, συγγνώμη, ε, αρχίζει η ψηφοφορία. 261 Τέλος εφορία Εγκρίνεται. 262 ψηφίζουμε τώρα. Εγκρίνεται λοιπόν. Πάμε στην τροπολογία της Επιτροπής Μεταφορών 15, δεύτερο τμήμα. Α, όχι, συγγνώμη. Πρώτα τη 263 πρέπει να ψηφίσουμε. 263. Εγκρίνεται. Και μετά και... Α, είναι μαζί αυτές. Μάλιστα. Λοιπόν, μεταφορές 15. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Ψηφίσατε όλοι. Συμβαστική 16 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 67. Σάλτερ Μόζες Σίμψον. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 της Επιτροπής Μεταφορών. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 270. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το 271, Λαβία και άλλοι. ...269... Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17... Εγκρίνεται. ...273 Σιλβέστρης. Εγκρίνεται. Τώρα την 64, Σαλντεμόζη και άλλων. Ψηφίζουμε. Εγώ θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Τραν 11. Εγκρίνεται. Ένβη 29. Απορρίπτεται. 28 ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. Γκίτλινγκ 2. 2. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 3. Τρεμόζα και άλλοι. Απορρίπτεται. Τέσσερα δελάγγε. Εκρίνεται. Συμβιβαστική ένα στο εκτιμώντας β. Εκρίνετε. Τροπολογία 15 τώρα, πατραων Νέβες. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 76 έραντς και άλλων. Θα έλεγα πως εγκρίνεται εγώ. Εγκρίνεται. Δεκάξι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17 στο Ιανοφ ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται, μου φαίνεται. Ναι, απορρίπτεται. 19. Εγκρίνεται. 26. Απορρίπτεται. Τριάντα. Σκοτά. Απορρίπτεται. 29. Απορρίπτεται. 27. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 31. 31 Ρέιμερς, τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 28 Dodge ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 32 για Απορρίπτεται. 34. Εγκρίνεται. Πάμε στην 24. Η Έγκλε. Εγκρίνεται. 25. Γκαρσία Περές. Απορρίπτεται. 36. Νταντά. Απορρίπτεται. 38. Βερσία και άλλη. 38 δεν έχει πλειοψηφία. 39. Ψηφίζουμε για τα 39. Απορρίπτεται. 40.

εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Εγκρίνεται. Pagina successiva, votiamo l'emendamento 57. Ε, περνάμε στη 57. 57 πατραονέβες. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 59. Ψηφίζουμε για την 59. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Τροπολογία ένα τελάγγε, Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στα ψηφίσματα. Αυτά δεν χρειάζεται να τα ψηφίσουμε γιατί καλύπτονται. Μένει μόνο η τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα αυτό όπως κοπήθηκε. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται λοιπόν. Τελειώσαμε με την έκθεση Βοζιχόφσκι. Συγχαρτήρια στον εισηγητή και ευχαριστούμε και τους συναδέλφους που ήταν εδώ για να ψηφίσουν. Και τώρα πάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση στους αυξανόμενους ε, κινδύνους ε, αντίστασης στα μικρόβια. Μάλλον μικροβίων. Αντίσταση των μικροβίων. Siamo tutti pronti. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Αρχίζουμε. Συμβιβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία για την πρώτη συμβαστική. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 4 τώρα. Υπέρ, ε, ε αρχής ψηφοφορία, συγγνώμη, πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη συμβαστική παριθμών 2, αρχής ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 τώρα. Ηλεκτρονικά πάλι. Την 8 πέρας εγκρίνεται. Η τροπολογία 9 αρχίζει ψηφοφορία. Τελειώνει. Εγκρίνεται. Η 10 ηλεκτρονική και πάλι αρχίζει. Κατά. Αποχέ. Αρχιποχέ, συγγνώμη, εγκρίνεται. Η συμβαστική 3 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και η συμβαστική παρελθόν 3. Ψηφίζουμε τη τροπολογία 14, αρχίζει η ψηφοφορία για τη 14. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει. Εγκρίνεται. 18 αρχίζει η ψηφοφορία. Γιατί 18 πέρας εγκρίνεται. 19 ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάλι αρχίζει. Πέρας εγκρίνεται. 20 αρχίζει η ψηφοφορία. Για την 20 πέρας εγκρίνεται. 21. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τελειώνει. 21 εγκρίνεται. Η τροπολογία 22. Σάρμπο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τελειώνει. Απορρίπτεται. 23. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τελειώνει για την 23. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την 24 Χόισλινγκ αρχής ψηφοφορία. Τελειώνει. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 4. Συμβιβαστική 4. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Ακολουθεί 28 ρόντου θα αρχίζει η ψηφοφορία. Τελειώνει. Απορρίπτεται. 29, αρχίζει η ψηφοφορία για την 29. Τελειώνει. Εγκρίνεται. Η 32 Σάρμπου αρχίζει η ψηφοφορία για την 32. Τελειώνει. Εγκρίνεται. 34 αρχίζει η ψηφοφορία. Γιατί η 34 τελειώνει. Εγκρίνεται. 35 ε, Νίκολσον αρχίζει η ψηφοφορία. Τελειώνει. Εγκρίνεται. Πάμε στη 40 τροπολογία. Πάντα το κυρίο Νίκολσον αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. Θα έλεγα, εγκρίνεται, ναι. Και τώρα θα ψηφίσουμε την 39 Aylward. Αρχίζει η ψηφοφορία, τελειώνει. Για να δούμε, εγκρίθηκε. Η 41. Αρχίζει η ψηφοφορία για τη 41 πέρας, νομίζω εγκρίνεται. Ναι. Ε, ψηφίζουμε τις 42 υπέρ συγγνώμη, αρχή ψηφοφορία. Τελειώνει. Εγκρίνεται. 43 αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τη 47. Ταντσίλα. Να ψηφίσατε όλοι. Πέρας, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε τη 48. 48. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 49. Σιλβέστρης. Αρχίζει η ψηφοφορία. Με τη 49. Πέρας. 49 εγκρίνεται. Η 50 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα, εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την 52. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 52. Πέρας. Εγκρίνεται θα έλεγα. Και τέλος το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε η τελική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται λοιπόν το σύνολο. Ευχαριστούμε τον Μάρτιν Χόισλινγκ. Μπράβο Μάρτιν. Και πάμε στο σημείο 6 τώρα. γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Βλέπω εδώ τον Λουίς Πάολο Άλβες, συγγνώμη. Όπως γνωρίζετε, εμείς είμαστε εδώ συνδεδεμένοι επιτροπή αυτή τη διαδικασία και έχουμε συναρμοδιότητα σε ό,τι αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3. Έχουμε συμφωνήσει με την αρμόδια Επιτροπή Απασχόλησης να ψηφίσουμε τη γνωμοδότησή μας στις 5 Νοεμβρίου και εκείνοι να μπορέσουν να ψηφίσουν στις 6 Νοεμβρίου. Για να γίνει αυτό η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είχε οριστεί για τη 12η Οκτωβρίου. Όπως σας έχει ήδη κοινοποιηθεί. Θα δώσω το λόγο στον ε, συντάκτη της γνωμοδότησης, τον Λουίς Παόλο Άλβες και βεβαίως στους εκπροσώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρίστανται και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Έχει το λόγο, Λουίς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα του αρχίσω να κάνω ένα προκατακτικό σχόλιο για την ίδια μου την παρουσίαση. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην προσπάθεια που έκανε η Επιτροπή Γεωργίας, ούτως ώστε να διαθέτει τις απαιτούμενες αρμοδιότητες και άρα τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τους γεωργούς στα πλαίσια αυτής της πρώτης κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσημα, ε, δια του Προέδρου της, ανέλαβε 7 πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η Επιτροπή Απασχόλησης και ε, η διάσκεψη των Προέδρων προσπάθησαν ε, να επιτύχουν αποκλειστική ή ενίοτε μεικτή αρμοδιότητα για τα άρθρα που έχουν κέρια σημασία, ούτω ώστε η Επιτροπή Γεωργίας να μπορέσει να ε, προστατεύσει τους γεωργούς, ξαναλέω, στο πλαίσιο αυτού του σχέδιου κανονισμού. Το άρθρο 4.3 ορίζει τα συγκεκριμένα κριτήρια που ισχύουν στο τομέα της γεωργίας Ζητάμε και αποκλειστική αρμοδιότητα. Επίσης, ο ορισμός καθώς και το πεδίο εφαρμογή όσον αφορά στη Γεωργία, άρθρο 23 για την διαχείριση των γεωργικών ταμείων, όλα τα άρθρα που ενέχουν τα ειδικά ε, χαρακτηριστικά της γεωργίας, για αυτά ζητάμε αποκλειστική αρμοδιότητα. Ξαναλέω για να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή μας να υπερασπιστεί τους γεωργούς ε, σε σχέση με αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πρωτοβουλίες αυτές σε διάστημα ενός έτους απερίφθησαν και γι' αυτό κάνω αυτήν την παρατήρηση. Φτάσαμε στο σημερινό στάδιο χωρίς καμία αποκλειστική αρμοδιότητα τελικά για αυτή την πρόταση. Η μοναδική αρμοδιότητα που καταφέραμε να αποκτήσουμε είναι μια ε, μεικτή αρμοδιότητα για το 4-3 σε σχέση με τις πράξεις κατεξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά ε, δεδομένου του διαλόγου στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, αυτή τη στιγμή μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι επιτροπές όπως αυτή της ανάπτυξης της υπαίθρου δεν μετέχουν στην όλη διαδικασία η Επιτροπή Απασχόλησης κατέθεσε πρόταση για να καταργηθεί ε, η πράξη κατεξουσιοδότηση εξουσιοδότηση αρμοδιότητα δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που έχουμε φτάσει δεν έχουμε καμία δυνατότητα να υπερασπιστούμε ειδικά συμφέροντα των γεωργών. Επίσης ε, με αυτή τη διαδικασία πράξης ε, κατεξουσιοδότηση βάσει της οποίας έχει λειτουργική δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπεραμεινθεί των συγκεκριμένων γεωργικών συμφερόντων αλλά επειδή δεν έχει καμία συγκεκριμένη μελλοντική προοπτική, θα χρησιμοποιηθεί η πράξη κατεξουσιοδότηση μόνο για αυτόν τον κανονισμό. Το αποτέλεσμα είναι ότι η έκθεση που τώρα σας παρουσιάζω ακολουθεί ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει και ένα διαφορετικό προσανατολισμό, εάν όμως ήταν διαφορετικό και το πλαίσιο και τα απεπραγμένα μέχρι στιγμής. Λοιπόν, τώρα θα σα εκθέσω την άποψή μετά από αυτή την πρώτη παρατήρηση. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση για την περίοδο 2014 2014-2020 έχει ως στόχο να προστατεύσει τους ε, εργαζομένους, ε, να ε, διευρύνει την κάλυψη στους ανεξάρτητους επαγγελματίες, καθώς και να προβλεθούν οι απαιτούμενες διατάξεις για να συμμορφωθούμε με τις διεθνείς ε, υποχρεώσεις μας. Αυτό είναι απαραίτητο για τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε την δυνατότητα διατήρησης αυτής της ενίσχυσης, κυρίως εν ώψη της κρίσης που βιώνουμε, αλλά και για μελλοντική χρήση. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία στο σχέδιο η πρόταση κανονισμού να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν, διότι ε, οι εργαζόμενοι ε, βρίσκονται αντιμέτωποι με ολέθριες ε, καταστάσεις και χρειάζονται βοήθεια. Είναι άνευ η κρίση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το πλαίσιο και λόγω των μεγάλων δυσκολιών είναι απαραίτητο να εγκριθεί το σχέδιο για το Ευρωπαϊκό αυτό ταμείο. Σε σχέση με τους συντελεστές συγχρηματοδότησης ε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα καποια κάποια κράτη-μέλη δεν δίνανται να χρησιμοποιήσουν σωστά αυτά τα ταμεία, όπως και για τα διαρθρωτικά ταμεία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο πρέπει να έχει ευνοϊκότερους συντελεστές για τις ε, πιο ευαίσθητες περιοχές για να επιτύχουμε τη σύγκληση για τις εξόχως απομακρυσμένες ή για τις ε, παράκτιες περιοχές, παραδείγματος χάρη. Ε, ήδη έχει εγκριθεί μια αρχή βάση της οποίας θα ευελτιωθεί η απορρόφηση από πλευράς ε, των κρατών μελών ε, που δέχονται εξωτερική ενίσχυση. Η οι διατάξει αυτέ προβλέπουν στον κανονισμό 11 του 2011. Χρειάζεται δηλαδή μια προσάυξηση τη τάξη του 10% όταν κάποια κράτη-μέλη, κάποιε περιοχέ προσφεύγουν στο Ταμείο. Βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει η πρόθεση να διευρυνθεί η κάλυψη και στους γεωργούς, ούτως ώστε να ε, αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών συμφωνιών και αναγνωρίζεται η, η αναγκαιότητα να δοθεί ιδιαίτερη δική σημασία στον τομέα της γεωργίας και των γεωργών και χρειάζεται πράξη κατεξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα έχει δυνατότητα παρέμβασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον ειδικό τρόπο που χρειάζεται στον τομέα αυτό βάσει και του κανονισμού που στόχο έχει να καλύψει τις ειδικέ ξαναλέω συνθήκες που ισχύουν στον τομέα της γεωργίας. Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε τους γεωργούς από τα αποτελέσματα των διεθνών εμπορικών συμφωνιών είναι ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταμείο. Γνωρίζουμε όμως ότι ε, θα μπορούσαμε να έχουμε γεωργού σε συγκεκριμένε παραγωγέ, συγκεκριμένε περιοχέ που χρειάζονται ειδική ενίσχυση, ούτω ώστε να μπορέσουν να προστατευτούν από τι ε, αρνητικέ επιπτώσει αυτών των συμφωνιών. Η Κομ Άγκρη ε, ε, αμφιβάλλει για την αποτελεσματικότητα αυτού του εργαλείου, αν δηλαδή μπορούν να δοθούν ικανοποιητικέ απαντήσει για του γεωργού με κάθε μέσο πάντως χρειάζεται η νομοθετική αρμόδιότητα ε, και η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μπορέσει να ε, προβεί στις απαιτούμενες ρυθμίσεις ειδικές για τους γεωργούς. Ε, η δυνατότητα παρέμβασής μας έχει αποδυναμωθεί και θα αποδυναμωθεί ότι περαιτέρω με την έγκριση του ε, σχεδίου κανονισμού πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η επικρατούσα θέση στην πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων και των ε, ε, επιμέρους επιτροπών είναι ε, η χρήση αυτή της πράξης σε κάθε εξουσιοδότηση και τη αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσει να ρυθμίζει αυτές τις ειδικέ περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα της πρότασης κανονισμού δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί στον τομέα της γεωργίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητικέ απαιτήσει για να καλυφθούν οι ειδικέ ανάγκε των γεωργών λόγω των αρνητικών επιπτώσεων διμερών και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών. Αυτές οι συμφωνίες ε, που επηρεάζουν ε, τη γεωργία ε, συνιστούν ένα δυσεπίλητο και λεπτό ζήτημα και το, η λύση θα ήταν να έχουμε ένα σχέδιο κανονισμού που να προβλέπει αυτή την αρμοδιότητα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλιστούν, ξαναλέω, ειδικέ απαντήσει για τι ανάγκε των γεωργών. Πέρα από την ιδιαιτερότητα αυτού του τομέα, τίθεται και το γενικότερο ζήτημα τη ε, μεταρρύθμιση ε, τη κοινή ε, γεωργική πολιτική. Γι' αυτό σα λέω ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή τη παρούσα πρόταση και να προσδώσουμε τα απαιτούμενα χρηματοπιστωτικά μέσα, ούτω ώστε στο πλαίσιο πλαίσιο του συνολικού προπολογισμού τη ΕΚΑΠ να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύψει τι ανάγκε των γεωργών. Γι' αυτό η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να προβούν στα απαιτούμενα διαβήματα για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Bene, grazie Alves, la situazione. Ωραία. Alves, όντω έτσι έχει κατάσταση όπω την περιέγραψε, Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη συζήτηση. Έχουν ζητήσει το λόγο ο Νικολέσκου και μετά ο Τζόρτζ Λάιον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και σας και τον εισηγητή και να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε. Για την Ευρωπαϊκή Γεωργία χρειαζόμαστε χρήματα και από τα προγράμματα της ανάπτυξης υπαίθρου και να έχουμε χρηστή διαχείριση και εξυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων. Δεν μπορούμε να λέμε ε, στους ε, αγρότες ότι θα τους βοηθήσουμε να κατεβάσουν τα ρολά για να βάλουν λουκέτο. Θα πρέπει να τους ε, βοηθήσουμε να ξεκολουθούν να είναι αγρότες. Και όταν ένα ταμείο ε, έχει αποδείξει ότι είναι αναποτελεσματικό, γιατί να το εφαρμόσουμε και στη Γεωργία, αφού υπάρχει ειδικό ταμείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεν καταλαβαίνω γιατί το προτείνεται αυτό. Ε, ο κύριος Λάιον. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Άλβες για τη ε, γνωμοδότηση, τις τροπολογίας και τη θέση που έχει λάβει. Εγώ ανέκαθεν θεωρούσα ότι οι προτάσεις για το Ταμείο για την Πακοσμιοποίηση ε, ήταν ε, πραγματικά άσκοπες και ε, μάλιστα και επιβλαβείς για τη Γεωργία. Καταρχάς, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο θα βοηθηθούν οι αγρότες από αυτό το ταμείο. Ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτά είναι επιπλέον χρήματα για τη Γεωργία. Αυτό είναι ανοησία, αφού έχει περιοριστεί η χρηματοδότηση του Ταμείου ε, συνολικά σε σχέση με την προγραμματική περίοδο 2007-2013, σε αυτό που προτείνουν για την επόμενη περίοδο 14 με 20. Είναι τελείως ανόητο αυτό που λέει ότι είναι έξτρα χρήματα για τη Γεωργία. Αφήστε που είναι υπόσχεση αυτή των κρατών μελών ότι κάποια στιγμή θα πληρώσουν. Δεν είναι κονδύλι του προπολογισμού. Εάν και εφόσον υπάρξουν οι ε, προϋποθέσεις και οι συνθήκες για τους αγρότες. Εγώ ανησυχώ πραγματικά. Δηλαδή να τάξουμε στους αγρότες ότι έχουμε ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουν την κρίση και μετά να μην τους τίποτα. Αυτή ήταν η πρώτη ανησυχία. Έχω και άλλη όμως. Ο Επίτροπος Εμπορίου τα έχει όλα αυτά ρυθμίσει. Υποτίθεται ε, προς όφελος ε, των αγροτών. Αντί να ασχολείται με τα θέματα εμπορίου όταν κάνει ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες εμπορικές, ασχολείται με τέτοια θέματα. Δηλαδή ο κίνδυνος να το δεχτούμε ποιος είναι επιτρέπουμε στον Επίτροπο Εμπορίου να επισέρχεται σε αυτά τα χωράφια και να κανονίζει τι θα κάνουν, ξέρω εγώ, οι βοοτρόφοι ή άλλη κατηγορία αγροτών και πώς θα ε, λαμβάνουν αντισταθμίσματα σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες. Θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ επιπόλαιο από πλευράς μας. Ε, είναι δούριο ύπος αυτό, ε, όπως σας είπα, είναι ένα τέχνασμα για να μας τη φέρουν. Για το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, η συγχρηματοδότηση για τη Γαλλία και την Ισπανία, για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειές τους, τις υπερπόντες, τα προγράμματα ΠΟΣΕΙ κτλ. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή αυτό. Πολλές τροπολογίες θα κάνω και εγώ και ελπίζω να τις εγκρίνουμε. E Πολύ ωραία. Ο Χόισλινγκ. Ευχαριστώ. Συνήθως δεν συμφωνώ με τους φιλελευθέρους, αλλά στο συγκεκριμένο υποστηρίζω απολύτως τον συνάδελφο. Και ευχαριστώ και τον συνάδελφο Άλβες για την γνωμοδότησή του. Ποιο είναι εδώ το αποφασιστικό. Τι πολιτικό μήνυμα θα στείλουμε. Και το πολιτικό μήνυμα είναι ότι Δεν συμφωνούμε με την ιδέα ότι με το ε, Ταμείο Παγκοσμιοποίησης μπορούμε σχετικά φθηνά να εξυπηρετήσουμε την ε, ε, υπόθεση των αγροτών. Ακούσαμε για τη Μερκοσούρ. Αν γίνει τέτοια εμπορική συμφωνία θα έχει τεράστιες συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και τώρα να έρθουμε με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης να κατευνάσουμε τους αγρότες, το θεωρώ και πλάνη. Και θα πρέπει να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, οι αγρότες δεν συμφωνούν και η Επιτροπή Γεωργίας. Θα πρέπει να υπάρξει άλλη αντιμετώπιση της Γεωργίας και σε σχέση με το Μερκοσούρ. Αυτό είναι ένα δηλητηριασμένο δώρο. Ε, δεν μπορούμε από εκεί να αντλήσουμε κονδύλια και να το εξηγήσουμε στον Επίτροπο Εμπορίου, να το καταλάβει ότι ε, είμαστε αδιαπραγμάτευτοι σε αυτό. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 3, ότι τα χρήματα αυτά είναι για τη γεωργία και να δούμε πώς θα τα ρυθμίσουμε. Αλλά το χρησιμοποιούν αυτό ως δελεάρ μας δίνουν 7 για να συμφωνήσουμε με εμπορικές συμφωνίες που δεν είναι συμφέρουσες για μας. Όχι. Ε, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτά, τώρα δεν ξέρω, ε, θα πρέπει να το δεχτούμε. Ε, και αυτά που λέγουν οι τροπολογίες είναι ο σωστός δρόμος, αλλά να το εξηγήσουμε με τόση σαφήνεια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι είμαστε στην Επιτροπή Γεωργίας όλοι ενωμένοι, θέλουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εμπορικών συμφωνιών και των επιπτώσεών τους στη Γεωργία. Και επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι το είπε και ο Λάιον, αυτά τα λεφτά που υπολογίζονται για τη Γεωργία, ότι κοιτάξτε, σας αναλογεί και από εκεί ένα μερίδιο, δεν ισχύει. Καταρχάς, δεν προορίζεται αυτό στη Γεωργία, ούτε πρόκειται να το πάρει η Γεωργία. Και μην νομίζουμε ότι έχουμε δισεκατομμύρια που θα δώσουμε τώρα στους αγρότες. Δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση η Γεωργία σε θέματα ε, εμπορικών συμφωνιών άλλο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Και στις ελεύθερες συμφωνίες έχουμε και άλλη άποψη, ε, ελευθέρων συναλλαγών ε, εννοώ, και για τη Μερκοσούρ πρέπει να υιοθετήσουμε τελείως διαφορετική τακτική και θα χαιρόμουν ως αρμόδια για τη Γεωργία Επιτροπή σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις αν μας συμπεριελάμβαναν και επί της ουσίας και όχι να έρθουμε να ευλογήσουμε το αποτέλεσμα δεν είναι συμπεριφορά αυτή ούτε τρόπος μεταχείρισης ενό τόσο σημαντικού θέματος. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Αντρέα. Θέλω να υπογραμμίσω όμως αυτό που είπε ο Μάρτιν, ότι η πόρα είναι της γεωργίας. Το είπε ο Επίτροπος και η Επίτροπη. Εμείς πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, γιατί η συζήτηση, στη... για να είναι μάλλον σαφή σε αυτή η πτυχή και στη συζήτηση μέσα στις ομάδες. Και όταν θα βρεθεί η στιγμή για τις δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να θυμίσουμε ότι πριν αγγίξουμε τα κονδύλια της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής υπάρχουν και άλλα κονδύλια. Ο Άντρε. Ο Άντρε, ε, ναι, ευχαριστώ. Νομίζω πως όντω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά αυτό, αυτό το Ταμείο παγκοσμιοποίηση. Και μάλιστα συμμερίζουμε σε μεγάλο βαθμό τα όσα είπε ο Λουίς θα πρέπει σε αυτή την πρόταση της Κομισιόν να δούμε την αντίφαση που υπάρχει. Να αποφύγουμε τι αρνητικέ επιπτώσει των εμπορικών συμφωνιών ε, επί τη Γεωργία. Άρα λοιπόν θα πρέπει διαφορετικά να διαπραγματευτούμε αυτέ τι συμφωνίε. Θα πρέπει καταρχήν να βγούμε από αυτή την προσέγγιση του απόλυτου ελευθέρου εμπορίου για τα γεωργικά προϊόντα και όπου η θέση τη Κομισιόν δεν είναι συνεκτική. Δηλαδή, από τη μια προωθεί την απελευθέρωση και στον τομέα τη Γεωργία και μετά αναγνωρίζει ότι οι συνέπειε είναι αρνητικέ. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν την πρόταση μεταφοράς των κονδυλίων στην κοινή γεωργική πολιτική. Εγώ θα ήμουν πολύ πολύ προσεκτικός γιατί η δουλειά που γίνεται για τις δημοσιονομικές προοπτικές δεν έχει ακόμα κλείσει. Ε, θα πρέπει να προσέξουμε μήπως αυτό το κονδύλι θα, μπορεί, θα μπορούσε να είναι συνοδευτικό, να μπορούμε να το μετρήσουμε και έπειτα θα πρέπει να φανταστούμε ότι αυτά αυτές οι πιστώσεις έρθουν στην κοινή γεωργική πολιτική ενώ τα κράτη-μέλη δεν έχουν εγκρίνει τον προπολογισμό. Μάλιστα, ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η Έστερ Εράνς Γαρσία και μετά ο Άλμπερτ Ντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε δεν ε, έχω αλλάξει άποψη ε, σε σχέση με τα όσα λέω τόσο καιρό και όσα ακούγονται και εδώ. Είναι υποσχέσεις και εικονικά χρήματα. Τώρα να βάλουμε ένα κεφάλαιο για τη γεωργία στο Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης για να ελπίζουμε ότι θα ε, αποζημιώσουμε γεωργούς και κτηνοτρόφους για τις συνέπειες από την, ε, τις εμπορικές συμφωνίες ε, εμένα μου φαίνεται ρηψοκίνδυνο ε, και αρκετά πεδαριώδες να αντιταχθούμε στην προσπάθεια αυτή. Γιατί τι κάνει το Συμβούλιο στις δημοσιονομικές προοπτικές, ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχουν κράτη-μέλη που θέλουν να συνεχίσουν να κόβουν από τη Γεωργία για να δώσουν λιγότερα στον προπολογισμό και δεν μου φαίνεται πολύ ρεαλιστικό να λέμε ότι ε, να μην έχει καθόλου χρηματοδότηση η Γεωργία από το Ταμείο ε, και θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αλλιώ. Ε, η απώλεια εισοδήματο των Γεωργών θα καλυφθεί από αλλού. Νομίζω ότι χρειάζεται μία πολυμέτωπη επίθεση εδώ και να δείξουμε και κάποια τακτική. Εγώ δεν θα απεμπολούσα σε καμία περίπτωση το γεωργικό κεφάλαιο μέχρι να ε, πετύχουμε αμοιβαιότητα στις διεθνείς συμφωνίες. Ούτε θα απεμπολούσα στο να υπάρξει κεφάλαιο για τη γεωργία στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ενώ δεν θα έχουμε ακόμα την ασφάλεια ότι θα υπάρξει μια κοινή γεωργική πολιτική στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Δεν θα το απεμπολούσα καθόλου σας είπα ότι είμαι η πρώτη που δεν πιστεύω στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, αλλά να πούμε τώρα όχι, σημαίνει ότι θα αφήσουμε να χαθεί μια ευκαιρία που μπορεί στο μέλλον ενδεχομένω να μας χρησιμεύσει. Ευχαριστώ. Sì, eh, do la parola ad Είναι προφανές ότι τα όσα είπε ο Λουίς Άλβες ότι η Επιτροπή Απασχόλησης θα αναιρέσει κάθε αναφορά στον Γιώργο. Είναι μια θέση ρεαλιστική. Είναι σαφές ότι είναι πολύ περίπλοκο να σκεφτούμε τη μεταφορά των χρημάτων, αλλά από το Ταμείο, από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης στην κοινή γεωργική πολιτική, αλλά είναι το ίδιο περίπλοκο να φανταστούμε ότι κατά κάποιο τρόπο θα υπάρχει εκεί μέσα κάποιο όφελος για τους γεωργούς. Το λόγο έχει ο Άλμπερτ και μετά ο Μισελ Νταντάν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή Λουίς Άλβες για τη γνωμοδότησή του, αλλά και τους συναδέλφους, γιατί ε, βλέπω ότι υπάρχει ευρύτατη ε, συμφωνία εδώ. Ο πρώην ε, Υπουργός Γεωργίας της Βαβαρίας, γνωσμένου κύρους προσωπικότητα και πολύ σημαντικό στη Γερμανία τότε, είχε πει το εξή σημαντικό η γεωργία δεν συγκρίνεται με άλλους κλάδους της οικονομίας. Δυστυχώς ο Επίτροπος Εμπορίου εδώ στις Βρυξέλλες δεν έχει πάρει μυρωδιά και θέλει να βάλει τη γεωργία σε αυτό το γενικό τσουβάλι. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Ε, την περασμένη θητεία, αν δεν απατώμε, στο Στρασβούργο είχαμε υποβάλει μια τροπολογία εγώ μαζί με 78 συναδέλφους και ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο με πάνω από δύο τρίτα πλειοψηφία και λέει εκεί περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς τι λέει, ότι οι γεωργικές εισαγωγές και εισαγωγές τροφίμων επιτρέπονται μόνο εφόσον έχουν τις ίδιες προδιαγραφές για το περιβάλλον, την υγιεινή, την προστασία των ζώων, την προστασία των καταναλωτών, κοινωνικές προδιαγραφές και τα συμπαρομαρτούντα. Να το θυμίσουμε αυτό στο ε, Επίτροπο Εμπορίου, αν δεν απατώ με ονομαστική ψηφοφορία πέρασε αυτό με 534 ψήφους. Δεν τα αντιλαμβάνεται αυτά Επίτροπος φαίνεται. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο αυτό της παγκοσμιοποίησης έχω την εντύπωση ότι είναι μαγική εικόνα και οπτική απάτη για να καθησυχάσουμε λίγο τους αγρότες ε, στην Ήπεθρο και τίποτα. Ούτε καν εικονικά χρήματα δεν είναι, ε, κυρία Εράνς. Ε, απλούστατα είναι οφθαλμαπάτη. Γιατί αυτό που πρέπει να αντισταθμιστούν σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν. Μπορεί να φτάνουν τα χρήματα για να τυπώσουμε μερικά έγγραφα, αλλά αυτές οι μαζικές ζημιές που θα υποστεί η Γεωργία δεν καλύπτονται με τίποτα. Έχεις δίκιο ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση, αλλά δεν νομίζω ότι εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτή η εμπορική συμφωνία πρέπει να προσέξουμε ε, ε, τι συνέπειες θα έχει στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ε, ψηφίσαμε για τις μεταφορές των ζώων. Έχω πάει στη Βραζιλία επανειλημμένα. Για να δούμε εκεί έτσι θα μεταφέρουν τα ζώα με τις, με τις δικές μας διατάξεις, με αυτά που ψηφίσαμε τώρα, τις ίδιες συνθήκες ακολουθούν στη μεταφορά των ζώων στη Βραζιλία. Και τώρα έχουμε και γεωργική μεταρρύθμιση. Θα πάει στο βρόντο ε, η γεωργική μεταρρύθμιση αν μετά πάμε και κάνουμε εμπορικέ συμφωνίες με γεωργικά κράτη. Να ξεχάσουμε τη γεωργία μας. Δεν θα έχει καμία προστασία. Δεν μιλώ για ποιοτική, καμία προστασία. Και τότε θα έχουμε προβλήματα και μπορούμε να το κλείσουμε το μαγαζί της Γεωργίας στην Ευρώπη. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μέσα σε αυτή την πρόταση ανάμεσα στα εργαλεία, τα μέσα που έχουμε και τις πιστώσεις. Ναι, χρειαζόμαστε ε, κονδύλια, πιστώσεις, ε, οι οποίες απορροφούνται από το κονδύλι για, τη γεωργία και πρέπει να εξευρεθούν μέσα στο, ε, στο συνολικό προϋπολογισμό ε, για τη μεταρρύθμιση κοινή γεωργικής πολιτικής στο συγκεκριμένο κονδύλι για αυτή τη δράση. Αλλά ε, για τα εργαλεία δεν χρειαζόμαστε νέα μέσα ουσιαστικά επανειλημμένα εδώ και στην Ολομέλεια σε θυελώδη συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε πει επανειλημμένα και πρέπει να το επαναλάβουμε ε, διότι φαίνεται ότι δεν κατέχει τη γεωργία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μπορούμε να αντικαθιστούμε εύκολα τις παραγωγές σε βιομηχανικό επίπεδο είναι όλα εύκολο για την ε, ε, νέα χρήση βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη υπάρχουν δυσκολίε. Αλλά ξέρετε, στον τομέα τη γεωργία, όταν κάποιε περιοχέ έχουν επιλέξει μία καλλιέργεια, σημαίνει ότι οι φυσικέ, κλιματικέ ε, και ε, εδαφικέ συνθήκε οδηγούν σε αυτήν την καλλιέργεια και δεν, με αυτά τα ψίχουλα αποκλείεται να επιτύχουμε αναδιάρθρωση. Τώρα, όταν ανοίγουμε την πόρτα για παραγωγές ε, που θα ε, ε, σκοτώσουν όλες τις παραδοσιακές καλλιέργειες της Ευρώπης δεν είναι ο ιδανικός δρόμος. Είδαμε και πριν από λίγους μήνες τη μελέτη για τον καπνό που παρουσιάστηκε εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας και δεν θυμάμαι που είδανε στη Βουλγαρία νομίζω ε, τέλος πάντων περιοχές που ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με αυτήν την καλλιέργεια και θυμηθείτε τι έλεγε η μελέτη ότι καμία άλλη καλλιέργεια μπορεί να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων απασχόληση, το ίδιο εισόδημα, την ίδια παραγωγή. Θυμηθείτε ε, με, τι έγινε με το Μερκοσούρα, αν, αν ανοίξουμε την αγορά μα στα κρέατα της Λατινικής Αμερικής, ε, ε, στην Γαλλία και στην Ιρλανδία υπάρχουν περιοχές που θα πέθαιναν. Πρέπει να καταδικάσουμε αυτό το μέσο που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να πούμε ναι στις πιστώσεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μισελ. Ο Αντιπρόεδρος Σικέρσκι και μετά θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν αν θέλει. Αναφέραμε εδώ στην Επιτροπή πολλές φορές ότι υπάρχουν ε, κάποιες διαφορετικές πτυχές σε αυτό το θέμα και ε, είναι συναρμοδιότητα διαφόρων επιτρόπων, όχι μόνο του κυρίου Τσιόλος. διότι είναι και ζήτημα προϋπολογισμού, είναι εμπορικό το ζήτημα, θα πρέπει παραδείγματος χάρη να ακούσουμε τον Επίτροπο αρμόδιο για τα εμπορικά ζητήματα να μας προβάλλει επιχειρήματα για να ενισχύσει τη θέση του ε, στο σώμα των επιτρόπων. Ε, αντικατέστησα τον πρόεδρό μας ε, ε, σε μια συνεδρίαση της διάσκεψης των πρόεδρων των επιτροπών. Συζητήθηκαν εκεί στρατηγικού χαρακτήρα ζητήματα που σχετίζονται με αυτή την πρόταση. Προγραμματίζαμε ταυτόχρονα και τις εργασίες μας ε, για το 2013. Και αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι γνωρίζει ότι με τις επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές ε, θα έχουμε αύξηση 12%. Δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει σε σχέση με τα νέα κράτη-μέλη και θα χρειαστεί να περιστύλουμε τις ε, πληρωμές προς κάποιες ε, χώρες ε, και σε περίοδο κρίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πιστώσεις, διότι είναι πολύ χαμηλά τα εισοδήματα. Είναι στα δύο τρίτα του μέσου εισοδήματος των άλλων χωρών. Γενικότερα όμως η Γεωργία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει ε, κρίση στον ε, τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και θα πρέπει να είμαστε πιο αγωνιστικοί, να είμαστε πιο επιθετικοί και να ε, υπερασπίσουμε τη γεωργία. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις από μακριά, τις εξελίξεις ενώ για το τον προϋπολογισμό. Πολλοί αγωνίζονται για τις αστικές και περιαστικές περιοχές και ε, παραγνωρίζουμε τη σημασία της γεωργίας. Όμως δεν είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Bene, grazie anche di Adesso darei la parola al direttore. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον... Μάρια Αρμεκίνες. Um, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ζητήσω το λόγο, γιατί φοβάμαι ότι βρισκόμαστε μεταξύ ε, σφύρας και άκμονος αυτή τη στιγμή. Θα, όμως είναι σημαντικό να απαντήσει η Κομισιόν ε, τα ερωτήματα του Μισελ Νταντέν και άλλων συναδελφών. Ε, δεν θέλουμε φυσικά τα χρήματα να φύγουν από τη Γεωργία, αλλά δεν θέλουμε αυτό να αποτελέσει μήνυμα ότι οι εμπορικές συμφωνίες είναι μια χαρά, γιατί υπάρχει κάποια στήριξη εκεί. Παρακαλώ λοιπόν να ακούσουμε την ε, Κομισιόν, όπως είπατε κιόλας. Molto Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Μαρία, για αυτή τη διευκρίνηση. Δίνω το λόγο να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Διευθυντή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Άλβες για την έκθεσή του, αλλά απαντήσω και στις ερωτήσεις. Για να εξηγήσω τι μας ενέπνευσε για τον κανονισμό αυτό το θέμα ε, για το μέσο και το θέμα της χρηματοδότησης του μέσου. Αρχίσω από τη χρηματοδότηση του μέσου. Τα ποσά αυτά πρόκειται να συζητηθούν στην οικοδόμηση, στην αρχιτεκτονική ολόκληρη του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό τον καιρό γίνονται συζητήσεις, αλλά το ταμείο αυτό είναι εκτός MFF, δεν είναι εντός του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ε, σε σχέση με τα ποσά που μπορούν να μεταφερθούν από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να συνεχίσω ε, τη συζήτηση ή την δικαιολόγηση και το πώς ε, έχει προβληματική του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και η δομή του. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, υπάρχει σήμερα και καλύπτει και ε, τους ε, ανέργους. Στο μέλλον, στη νέα πρόταση, καλύπτεται καλύτερα ε, γιατί μπαίνει σε αυτό το μέσο και μια άλλη κατηγορία, οι αγρότες. Κοιτούμε τι Οφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε από το μέσο αυτό, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής και τους δικαιούχους. Δηλαδή, δεν καλύπτουμε μόνο τους ανέργους γενικά, αλλά και τους ανέργους γεωργούς και κάποιους γεωργούς με κάποιες δράσεις για να μπορούν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Όταν βρίσκονται σε μια περιφέρεια ή σε ένα τομέα, υποπίεση και δύσκολες ε, περιστάσεις ως απόρρια μιας εμπορικής συμφωνίας ή ε, διάνοιξης του εμπορίου που θα μπορούσε ενδεχομένως θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες δυσκολίες για τους αγρότες. Πρόεδρε, δεν ήρθα εδώ για να συζητήσω τις συνέπειες και τα αποτελέσματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις γίνονται ξεχωριστά με τη δική σας βεβαίως συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια εμπορικών συμφωνιών. Και υπάρχουν συνέπειες από τις εμπορικές συμφωνίες που ενδεχομένως να δημιουργήσουν δυσκολίες και δυσχέρειες σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις για τους γεωργούς. Δηλαδή το συγκεκριμένο μέσο δίνει τη δυνατότητα να ε, δρομολογούνται κάποιοι μηχανισμοί ε, που θα υποστηρίζουν τους αγρότες ε, σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Όταν μπορεί κανείς εκ των προτέρων να κάνει ανάλυση των επιπτώσεων μιας τέτοιας συμφωνίας. Τίθεται τώρα το ερώτημα. Εάν βγει τελείως από το μέσο αυτό η Γεωργία, το μέσο παραμένει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την ε, Παγκοσμιοποίηση, για ε, κοινωνικές ρυθμίσεις. Αν κοιτάξουμε την τροπολογία υπαριθμών 3, τι λέει. Ότι θα είναι χειρότερο το σενάριο για τη Γεωργία, διότι ε, αποκλείονται απολύτως από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Αν παραμείνει το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, και σημειώνω τη δική σας γνώμη και με μεγάλη προσοχή, ε, αν ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση, θα αποκλειστούν οι αγρότες από το Ταμείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταργηθεί το Ταμείο. Και το Ταμείο θα υπάρχει και χρήματα θα ζητάει. Δηλαδή, ε, η ιδέα να μεταφερθούν πιστώσεις υπέρ των γεωργών στο παρόν στάδιο είναι κάτι ε, που το θεωρώ θετικό. Ξέρω ότι η πρόταση μιλά για 2,5 δις σήμερα από τα τρία που προβλέπονται για τη Γεωργία. Σημειώνω ότι αν εξαιρεθεί η γεωργία, το μέσο παραμένει, οι αγρότες είναι απ' έξω, δεν περιλαμβάνονται, γίνονται εμπορικέ συμφωνίες, ακολουθούν το δρόμο τους, ε, κάποια στιγμή θα ολοκληρωθούν και τι γίνεται, ένα μέσο που υπάρχει και ε, καλύπτει τουλάχιστον 12% σήμερα ε, των γεωργών, αύριο θα καλύπτει 0% αν τους εξαιρέσουμε και περάσει η τροπολογία 3. Οπότε, Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε, να δούμε πώς. Ε, ίσως χρειάζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση ε, το μέσο αυτό, το ταμείο για να εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό του, αλλά να μην καταργήσουμε κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, με επιτυχία. Θυμάμαι ότι είχαμε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης για ειδικέ περιστάσεις που θα τις έχουμε ε, ορίσει και να μην θεωρείται αντισταθμιστικός μηχανισμός για τους αγρότες. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο ε, στόχος είναι να υπάρξει μια ελάχιστη ενίσχυση τα έχουμε ταμεία για την ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά δεν απαντούν ε, σε αυτές τις δράσεις που προβλέπονται. Και ποιες είναι αυτές. Να σας δώσω παράδειγμα. βοήθεια, παροχή συμβουλών ε, για τον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων, για την απασχόληση. Είναι μια σειρά από δράσεις ε, που καλύπτουν το 90% ε, από αυτόν τον συγκεκριμένο μηχανισμό. Και αυτό πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτείται από το Ταμείο ε, Ανάπτυξης της Υπέρου. Ε, της Υπέθρου. Δηλαδή... Κάνουμε ένα άλμα από μια δομή που σήμερα υπάρχει σε μια άλλη που δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση για να λειτουργήσει. είναι πολιτική απασχόληση. Ωραία. Αλλά θα πρέπει να μπουν αυτά τα χρήματα στην κοινή γεωργική πολιτική, λέτε. Αλλά όπω σας είπα, οι συζητήσει για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αλλά δεν θα είναι εύκολο να βρεθούν κονδύλια για τη γεωργία. Γι' αυτό σας λέω και επιτρέψτε μου ότι βλέπουμε συμπάθεια εκείνου που λέγουν μην παρεξηγείτε το μέσο αυτό και τη χρηματοδότηση και μην χάσετε κάτι που υπάρχει από ένα εικονικό υποτιθέμενο σενάριο που μπορεί ποτέ να μην υλοποιηθεί. Γιατί θα υπάρξουν εμπορικέ συμφωνίε, θα υπάρξουν συνέπειε για του αγρότε και τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Α φροντίσουμε να υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για να αποφύγουμε δύσκολε καταστάσει. Αλλά εάν αύριο η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια που θα θα ε, ασκήσει πίεση σε κάποιους τομείς της γεωργίας, τότε ας μην χάσουμε ένα μέσο που υπάρχει και που μπορεί να βοηθήσει. Με συγκεκριμένη λύση, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα ε, και των αγροτών, γιατί είναι ταμείο έκτακτης ανάγκης σε ιδιαίτερες περιστάσεις. Ξέρω, Πρόεδρε, ότι λέγοντας αυτά, Υποστηρίζω βέβαια στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συγκεκριμένες δράσεις και όχι ένα γενικότερο πλαίσιο, ένα γενικότερο πεδίο που δεν βλέπω και πώς αυτό θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Sì, noi ringraziamo l'intervento della Commissione, ringraziamo il direttore. Ε, να ευχαριστήσουμε τον Γενικό Διευθύντη για την παρέμβασή του. Θα ήθελα όμως να σημειωθεί και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή Άλβες τώρα, σε λιγάκι. Ήθελα μόνο να πω ότι δεν είμαστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Η Επιτροπή Απασχόλησης είναι βασικά αρμόδια ε, επιτροπή και εκείνη ε, ω εκ τούτου δίνει τον προσανατολισμό, τον προσανατολισμό απόρριψης της θέσης αυτής. Καταλαβαίνουμε αυτά που λέτε, αλλά η πρότασή μας είναι προκλητική, η πρόταση δηλαδή του εισηγήτη. Θέλαμε να πούμε μόνο ότι πρέπει να βρεθούν και τα απαιτούμενα μέσα. Οπότε θα, ήθελα η Κομισιόν να πει τα ίδια πράγματα που, θα, που, θα, που είπε εδώ, όταν στις 6 Νοεμβρίου θα ψηφίσουν και στην Επιτροπή Απασχόλησης και θα ψηφίσουν με βάση τις ενδείξεις που μας έχουν δώσει μέχρι τώρα. Ε, πάντως ευχαριστώ την Κομισιόν και το λόγο έχει ο Λουίς Παόλο Άλβες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ έχουμε ένα θέμα ε, που δεν είναι αν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα ή αν χρειαζόμαστε μέσα για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της ε, παγκοσμιοποίησης ή τις ενδεχόμενες ε, συνέπειες αυτής. Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό λοιπόν που το, θέμα, το ερώτημα που τίθεται είναι υπάρχει ένας κανονισμός. Έχουμε και ένα ταμείο το οποίο και μάλιστα ήρθε από την Κομισιόν μια πρόταση κανονισμού, όπως είπε και ο Πρόεδρος, που η αρμοδιότητα δεν είναι της δικής μας Επιτροπής. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ε, με ποια μορφή αυτός ο κανονισμός, όταν θα εγκριθεί, θα μπορεί να υπερασπιστεί αυτά τα οποία πρέπει να υπερασπιστεί, δηλαδή τα συμφέροντα των γεωργών. Όπως είπε πολύ καλά ο Τζορ Λάιον, έχουμε φτάσει στο τέλος με μια γραμμή του προπολογισμού, αλλά χωρίς τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο, στο ταμείο. Πώς λοιπόν η ίδια η Κομισιόν θα παρεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία αν δεν υπάρχει νομική πράξη. Ε, σε αυτή την πρόταση είναι σημαντική η εκ των προτέρων έγκριση, ώστε να μπορούμε να ενεργήσουμε ακριβώς τη στιγμή που υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά το στοιχείο αυτό έχει χαθεί. Η ίδια η Κομισιόν δεν θα έχει κανένα τρόπο να παρέμβει στο Ταμείο και να εξυπηρετήσει την Γεωργία. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να δουλέψουμε όχι πια στο στο θεωρητικό επίπεδο. Θέλουμε να προχωρήσουμε, ε, να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα βήμα ως Κοινοβούλιο. Σε αυτή τη φάση η Κομισιόν δεν έχει νομικό εργαλείο στη διάθεσή της και αυτό χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε από εδώ και μπρος. Και το ερώτημα είναι, αξίζει τον κόπο να ε, εξασφαλίσουμε έναν κανονισμό που λέει ότι θα ε, τηρεί την ισότητα της μεταχείρισης. Αλλά αυτό δεν είναι το να μεταχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο αυτά που είναι ίδια και διαφορετικά αυτά που είναι διαφορετικά, γιατί η περίπτωση των γεωργών είναι διαφορετική για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Αυτό δεν θα συμβεί με αυτόν τον κανονισμό. Και εφόσον δεν θα συμβεί, δεν θα έχουμε τις απαραίτητες απαντήσεις. Ε, αυτό είναι το βασικό ερώτημα και δεν έχουμε απάντηση. Αν κάνουμε ένα βήμα εδώ, θα κάνουμε ένα βήμα προς τον κρεμό. Γιατί, Γεωργή, σε θέματα διεθνούς εμπορίου, εάν δεν τους υποστηρίξουμε, εάν δεν τους υπερασπιστούμε, εάν δεν έχουν πραγματικά μέσα στη διάθεσή τους, στα οποία όμως να έχουν πρόσβαση, και θα κάνουν πάνε ίσια για τον κρεμό. Είναι ένα βήμα το οποίο μετά δεν θα μπορεί να προσαρμοστεί. Πώς θα ανταγωνιστούμε ισότιμα με τους άλλους. Οι άλλοι χρειάζονται 500 αποστολές, 500 αγροκτήματα. Μα πώ θα είναι η δικιά μας γεωργία, τι σχέση έχει αυτό με τη δικιά μας γεωργία. εμεί χρειαζόμαστε ευαισθησία. Είναι ναι και η γεωργία εργαζόμενη, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι φυσιολογικοί αλλά η πρόταση αυτή από το μέσο πρόσβαση στο κονδύλι δεν είναι το καταλληλότερο υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτό είναι το ζήτημα και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αν θέλει να το αντιμετωπίσει και το Συμβούλιο, αν θέλει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες των γεωργών θα πρέπει να φτιάξει άλλο εργαλείο, άλλο μέσο. Γιατί όταν αυτό το μέσο εγκριθεί εδώ στο Κοινοβούλιο δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν γεωργό ώστε να αντέξει αυτές τις συνέπειες. Άρα δεν μπορούμε εδώ σε αυτή την Επιτροπή να θεωρήσουμε πως είναι ένα μέσο το οποίο να μπορούμε εμείς να επικαλεστούμε σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, γιατί είναι ένα μέσο το οποίο οι Γεωργοί δεν θα μπορέσουν ποτέ να το χρησιμοποιήσουν. Δεν συμφωνώ και δεν συμμερίζομαι λοιπόν την άποψή σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρα τα πράγματα και μπορούμε να κλείσουμε εδώ αυτή τη συζήτηση. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 12 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, γιατί πρέπει να ψηφίσουμε στις 5 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους και τώρα διακόπτουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής μας που θα συνεχιστεί το απόγευμα για να κάνουμε συνεδρίαση των συντονιστών για λίγα λεπτά ακόμα παρακαλώ να μείνετε εδώ. Θα έχουμε μια σύντομη συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ για τους υπόλοιπους. Θα τα πούμε στις 3.